αφορά ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά με τη μαζική κλίμαξα οργανωμένη κατασκοπή εκ μέρους της NSA και με εμπλοκή της Bundesnachrichtendienst εις βάρος πολιτικών και εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα δώσω το λόγο καταρχάς στην Επίτροπο την κυρία Γεωρόβα. Uh, Κυρίες και κύριοι, πάρα πολύ θετική ευκαιρία που σήμερα μας δίνεται να δούμε για το ποια είναι ε, αυτή η υπόθεση της συνεργασίας ε, όπως έχει δημοσιευτεί παντού μεταξύ ε, της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Αμερικής και της Γερμανικής. Σύμφωνα με τον έντυπο τύπο πάρα πολλά στοιχεία εδώ πέρα έχουν μείνει ασαφή. Πρώτα-πρώτα μέχρι ποιο βαθμού η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών έχει εμπλακεί Επίση, τι κατασκοπή έγινε από πλευρά τη NSA στην ε, Δυτική Ευρώπη βάρο κάποιων εταιριών ει παραβίαση του γερμανικού δικαίου. Γιατί αυτέ οι εταιρείε ε, εξασφαλίζουν την εθνική ασφάλεια και όλα αυτά είναι φεύγα θέμα ε, αποκλειστικά εθνική αρμοδιότητα. Δεν έχουν να κάνουν με το κοινωτικό δίκαιο ούτε με τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων αφορά μόνο τα κράτη-μέλη όταν εφαρμόζουν κοινωτικό δίκαιο. Πέραν τούτου, η έννοια της εθνικής ασφαλείας θα πρέπει πάρα πολύ στενά να ερμηνευθεί όταν χρησιμοποιείται από ένα κράτος μέλος για να επικαλεστεί το μη εφαρμόσιμο του κοινοτικού δικαίου. Και το Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων λέει ότι για να υποστηριχθούν τέτοια επιχειρήματα, δηλαδή το να μην ε, ε, εφαρμόσει το κοινωνικό δίκαιο θα, θα, πρέπει αυτό να αποδειχθεί και όχι απλώς να το επικαλεστεί το κράτος μέλος. Άρα θα πρέπει να δούμε τι γίνεται για τις ε, σχέσεις μεταξύ υπηρεσία πληροφοριών και μιας τρίτης χώρας. Αυτό είναι θέμα εθνικό και το κράτος μέλος θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει και αυτό θα γίνει ε, επί τη βάση τη εθνική νομοθεσία και στα πλαίσια της Σύμβασης Εθνικών ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Ε, ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει για πρώτος ομιλητή, ο κύριος Φω για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Το Σπίγκελ γράφει αυτή την εβδομάδα ότι το NSA προφανώς με τη γνώση της γερμανικής υπηρεσίας, ε, της μυστικής υπηρεσίας ε, παρακολουθούσε τμήματα της θετική Ευρώπης. Αυτό αποτελεί μόνο αυτά που γράφει η εφημερίδα. Δεν υπάρχουν ακόμα γνωστά. Δεν είναι ακόμα γνωστό το τι έχει γίνει. Τι συζητάμε, ότι οι μυστικές υπηρεσίες κάνουν αυτό που κάνουν. Μια ευρωπαϊκή υπηρεσία υποστήριξε ενδεχομένω μια άλλη φιλικά προσκύμενη υπηρεσία. Είναι καλό να διασφαλίζουμε ότι Υπάρχει τοποθέτηση από πλευρά μα σε ό,τι αφορά τη μαζική κατασκοπία και σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση πολιτικών, πολιτών και επιχειρήσεων ότι δεν τα αποδεχόμαστε αυτά. Αλλά αυτό το έχουμε διαπιστώσει ήδη. Γι' αυτό πιστεύω ότι η χρονική συγκυρία αυτή τη συζήτηση δεν είναι σωστή. Είναι πάρα πολύ νωρί και είναι και λανθασμένη και η τοποθεσία για να γίνει αυτή η συζήτηση. Δεν είμαστε το αρμόδιο μέρος για να κάνουμε τη συζήτηση αυτή. Θα πρέπει να φροντίσουμε να μην ε, δίνουμε την ψευδέστηση στους πολίτες ότι μπορούμε κάτι να επηρεάσουμε από εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν έχουμε τέτοια αρμοδιότητα για τις μυστικές υπηρεσίες, πόσο μάλλον για τις εθνικές μυστικές υπηρεσίες. Δεν έχουμε επιβεβαιωμένα γεγονότα. Γι' αυτό πιστεύω ότι αυτή η συζήτηση στο πλαίσιο εικασιών και υποθέσεων δεν είναι σωστή. Δεν υπάρχει ως τώρα υπόδειξη ή απόδειξη μαζικής κατασκοπίας, ούτε ενδοευρωπαϊκής κατασκοπίας και παρακολουθήσης. Όπως πάντα μιλάμε για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ περιοχών κρίσης και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε ίσως καλύτερα το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον έλεγχο των μυστικών υπηρεσιών. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά λέει τώρα η Πρόεδρος. Το λόγο έχει η κυρία Σίπελ. Ευχαριστώ και επιτρέψτε μου να κάνω μία πρώτη παρατηρήση. Δεν υπήρχαν μόνο ειδήσει στις εφημερίδες αλλά και τα μέλη του NSA και μέλη της δικής σας ομάδας και του δικού σας κόμματος ε, ε, επιβεβαίωσαν τα περιστατικά αυτά. Αλλά οι αποκαλύψεις ε, στα κράτη-μέλη δείχνει έχουν μείνει χωρίς ένα αφήσουν ίχνη και συνεχίζονται οι παρακολουθήσεις. Το Κοινοβούλιο όχι, όχι μόνο επικρίνει τη ΣΥΠΑ, αλλά έχει ζητήσει από τα κράτη-μέλη να ελέγχουν καλύτερα την κατασκοπία και να μην υπάρχουν περιπτώσεις μαστικής κατακτοσκοπίας. Και οι Βρετανικές και οι Γερμανικές μαστικές υπηρεσίες κατανομάστηκαν γιατί υπήρχαν εικασίες ότι δεν πήγαιναν τα πράγματα καλά εκεί. Δεν έχουμε ακόμα όλα τα γεγονότα επιτάπητος και σωστό. Αλλά θα δούμε πώς τοποθετούμαστε, πώς τοποθετούνται τα μέλη της Επιτροπής σε τέτοια σοβαρά περιστατικά. Όλοι ξέρουμε ότι όποιος ξεπερνάει τις αρμοδιότητες του, αν δεν είναι γνωστό ότι υπερβαίνονται οι αρμοδιότητες αυτές, είναι πραγματικά τρομακτικό αυτό, γιατί σημαίνει ότι δεν λειτουργήσε ο κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η μοναδική σωστή αντίδραση λοιπόν τώρα είναι ε, εκτεταμένη μελέτη έρευνα των όσων έγιναν από την Γερμανική Διερευνητική Επιτροπή και θα πρέπει εδώ να υποστηρίξουμε την έρευνα αυτή από πλευρά των κρατών. Ιδιαίτερο ρόλο δε παίζουν οι επιλογές όπως ε, ονομάζονται τους οποίους ήθελε να έχει η NSA για διάφορους σκοπούς. Και κλείνοντας να πω, φαίνεται ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να ασχολείται με το θέμα αυτό. Αυτό καταδεικνύει και η νέα νομοθεσία στη Γαλλία η οποία ε, δείχνει ένα γαλλικό Patriot Act. Θα πρέπει να συνεχιστεί σίγουρα η συζήτηση. Η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Επόμενη, ο επόμενος ομιλητής, ο κύριος Κρασνοντόφσκι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα αυτό πρέπει να πω ότι πιστεύω ότι η προλαλήσασα προσπάθησε να αντιμετωπίσει το θέμα με δίκιο τρόπο. Ή είπε ότι δεν είναι θέμα γερμανο-γερμανικό αυτό το ζήτημα. Γερμανός εκπρόσωπος ξεκίνησε τη συζήτηση αλλά δεν πρόκειται απλώς περί διαβιβάσεως πληροφοριών από την BND αφορώντας τους, που αφορούσε τους Ευρωπαίους πολιτικούς. Η κυρία Επίτροπος διευκρίνησε ότι επρόκειτο για τη Δυτική Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι επρόκειτο για όλη την Ευρώπη που αφορά το πρόβλημα και όχι μόνο τη συνεργασία με την NSA. Σε πολλά από τα άθρα στον τύπο τονίζεται το πρόβλημα που αφορά την υπηρεσία τη γερμανική, την 5, που συλλέγει Εβραίους πληροφορίες για τους πολίτες και τους πολιτικούς χωρίς να υπάρχει επαρκής δημοκρατικός έλεγχος. Σαν βουλευτής και πολίτης διαμαρτύρομαι λοιπόν γι' αυτό. Ολοκλήσατε τον χρόνο σας. Η κυρία Ιντεφελτ έχει το λόγο για δύο λεπτά τώρα, λέει πρόεδρο, αφού διέκοψε τον προηγούμενο μιλητή. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Πόσε φορέ έχουμε βρεθεί εδώ και να κουβεντιάζουμε παράνομη παρακολούθηση, κατασκοπία κατά των πολιτών, κατασκοπία κατά των πολιτικών, κατά των δημοσιογράφων, παρενόχληση των πληροφοριοδοτών. Μπορώ να επαναλάβουμε όλα τα, τα tweet, NSA, Belgacom, Τζαμάλτο, ε, κύριε Βος. Θα είχατε φυσικάσει τόσο πολύ αν δεν είχαμε μιλήσει για τις μυστικές υπηρεσίες, αλλά μιλούσαμε για τις κινέζικες υπηρεσίες. Και τι θα λέγαμε, αυτή είναι η δουλειά των μυστικών υπηρεσιών, κατασκοπεύουν. Ξεπεράστε το. Κοιτάξτε, εδώ έχουμε κανόνε στην Ήπειρο αυτή. Ποιο προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών μα. Ποιο θα προστατεύσει την ιδιωτική ζωή των πολιτών μα κύριε Βό. Σαφώς το ΕΛΚ δεν νοιάζεται καθόλου. Ούτε για την ιδιωτική μα ζωή, ούτε για το κράτο δικαίου, ούτε για το εθνές δίκαιο. Οι πολίτε δεν πρέπει να περιμένουν η αδίποτε προστασία από την πλευρά σα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα λέει ότι είναι αποκριστική αρμοδιότητα των κρατών μελών και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά σημειώνω το Συμβούλιο ξανά λάμπει για τι απουσίε του. Διότι αν είναι κάποιο θεσμικό όργανο που δεν δίνει, πώ να το πω, θα χρησιμοποιούσα κάποιο περίεργη λέξη που δεν νοιάζεται πολύ για τα δικαιώματα των πολιτών, αυτό είναι το Συμβούλιο. Αλλά κάποιο πρέπει να το κάνει αυτό. Και εγώ αρνούμαι να δεχτώ ότι όλα αυτά είναι νόμιμα και αποδεκτά. Πότε επιτέλους θα πάρουμε κάποιες απαντήσεις. Διότι αν αυτό μας κάνουν φιλικές χώρες, σκεφτείτε τι κάνουν οι χώρες που δεν είναι φιλικές για μας. Ο κύριος Βος είπε ότι δεν έχουμε αποδείξεις. Ε, βέβαια δεν έχουμε αποδείξεις. Ε, Λέγονται μυστικές υπηρεσίες για κάποιο λόγο, διότι αυτό που κάνουν είναι μυστικό. Γι' αυτό έχουμε έλεγχο κύριε Βος. Ο κύριος Βος δεν ακούει. Χρειαζόμαστε έλεγχο κατεπηγόντως εποπτεία, ευρωπαϊκούς κανόνες που θα εφαρμόζονται στις συνοριακές δραστηριότητες των μυστικών υπηρεσιών, διότι πρέπει να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό η κυρία Ernst έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ αυτό που το φανταζόμασταν πάντα ουσιαστικά αποκαλύφθηκε ότι όλες οι μυστικές υπηρεσίες, ακόμα και η γερμανική μυστική υπηρεσία, ε, τα κάνουν πλακάκια με την NSA, με φιλικές αρχές πάντα. Και οι κυβερνήσεις ε, όλες το ξέρουν. Οι Ευρωπαίοι πολίτες κλείνουν τα μάτια. Οι επιχειρήσεις παρακολουθούνται ε, οικονομική κατασκοπία σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό δίκαιο, με το εθνικό δίκαιο απαγορεύεται. Μα τι άλλο περιμένετε να γίνει δηλαδή. Μιλάμε για τους Αμερικανούς, για τους εκλογείς, για τη Γερμανία. Για την τέτοια χορήγηση πληροφοριών. Όλοι τα ξέρουμε τα περιστατικά αυτά και τα συζητήσαμε για το NSA. Οι μυστικές υπηρεσίες κάπου είχαν κάτσει και τα συζητούσαν και τρέβαν τα χέρια τους. Αυτή ήταν η αλήθεια την οποία πρέπει να συζητήσουμε. Δεν είναι μονομένη περίπτωση, δεν είναι μόνο η NSA. Είναι ένα σύστημα, ένα σύστημα ε, κατά παρακολουθήσεις εκατομμυρίων πολιτών, επιχειρήσεων, και σε κάποιες περιπτώσεις αυτό ονομάζεται έσχατη προσδοσία κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι ο λογαριασμό για τι επιστικέ υπηρεσίε που κάνουν ό,τι θέλουν και οι κυβερνήσει θα κρύβουν τα σκάνδαλα αυτά. Πόσο θέλουμε να τα, να τα υποστούμε όλα αυτά, να αφήσουμε αυτή την απάτη να συμβαίνει. Πιστεύω ότι θα πρέπει να μπει ένα τέλο λοιπόν σε αυτά. Thank ευχαριστώ. Για 1,5 λεπτό ο κύριος Άλμπεκτ. Thank you, President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητή Επιτροπή. Αν αυτές οι εκθέσεις του τύπου αποδειχτούν αληθινές, αυτό θα δώσει μια καινούργια διάσταση στο σκάνδαλο αυτό, που θα καταδείξει ότι το θέμα δεν είναι μόνο η NSA, η αλλά και οι δικές μας μυστικές υπηρεσίες, που δεν συνάδουν με τα πρότυπά μας, με τα θεμελιώδη δικαιώματα, με το κράτος δικαίου και τις αξίες μας. Και θα πρέπει να πω αξιότιμη επιτροπέ Γιούροβα ότι τώρα είναι η στιγμή να κάνουμε κάτι για την έρευνα αυτή. Αν ο όρος εθνικής ασφάλειας στην ε, συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, δεν τηρείται από τα κρατημέλη. Γιατί προφανώς αυτό συμβαίνει. Γιατί όταν αποκαλύφθηκε η υπόθεση Σνόντεν, η Άγγελα Μέρικαλ, είπε ότι η κατασκοπία σε φίλους είναι κάτι το οποίο δεν γίνεται. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι φίλοι της Γερμανίας ή να πούμε ότι δεν εννοεί τα λόγια της, δεν τα παίρνει στα σοβαρά τα ίδια της τα λόγια και νομίζω ότι αυτό είναι το θέμα για όλους τους ε, αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Θα πρέπει το Κοινοβούλιο να ζητήσει από τα κράτη-μέλη να πληρούν και να ανταποκρίνονται στα πρότυπα για την εθνική ασφάλεια και να ξέρουν ότι δεν κάνουμε κατασκοπία στο εσωτερικό της Ένωσης, γιατί υπάρχει ο χάρτης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα πρέπει να ανταποκριθούμε και να σεβαστούμε τις δικλείδες που προβλέπει η συνθήκη. Μάλιστα, τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Λεπρετό. Merci, Madame la Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Από το 2001 οι γερμανικές μυστικές επιχειρήσεις κατασκοπεύουν εταιρείε αλλά και προσωπικότητες και Γάλλους για λογαριασμό των ΙΠΑ και είχαμε αυτή την πληροφορία που προέρχεται από το Der Spiegel. Το επιβεβαίωσε η κυρία Μέρκελ και η καγκελάριος προσπάθησε να αρνηθεί τις ευθύνες της και κατηγόρησε τις μυστικές υπηρεσίες και είπε ότι πρόκειται για κάποιες αδυναμίες ε, τεχνικές και οργανωτικές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό. Ε, αποδεικνύει ότι μας έχει προδώσει η Γερμανία. Η, πρόδωσε το τον Ευρωπαίο τέρο της υπέρ των Αμερικανών. Επομένως χειραγωγούν οι Γερμανοί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά για να ωφελήσουν ε, τους Αμερικανούς και τα συμφέροντά τους. Άρα θα πρέπει να δούμε τις συνέπειες, να δούμε τι θα γίνει ε, και με το TTIP. Σα ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Για ένα μισή λεπτό. Ο κύριο Σιμπέρ. Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα σκάνδαλο κατασκοπίας. Σχετίζεται με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών των ήπα. Αυτό όμως ε, μας είχε υποσχοληθεί και στο παρελθόν. Άρα σήμερα δεν θα έπρεπε να μας υποσχολεί πάλι. Θα έπρεπε να μιλούμε για ασφάλεια. Όσοι δεν θέλουν να συζητήσουν κάτι τέτοιο, ισχυρίστηκαν ότι υπήρχε εδώ μυστική συνεργασία των υπηρεσιών πληροφοριών Γερμανίας και ΕΠΑ. Ε, βέβαια και αυτό γίνεται κρυφά. Πρόκειται για μυστικές υπηρεσίες πληροφοριών. Θα πρέπει να υπάρχει όμω τελικά για ποιου έλεγχο, γιατί εδώ διακυβεύεται η ασφάλειά μα. Η προστασία των δεδομένων είναι βασικό δικαίωμα το οποίο έχουμε ω φυσικά πρόσωπα. Θα πρέπει κάτι να γίνει γι' αυτό και θα πρέπει να προσαρμόσουμε και να επικαιροποιήσουμε τον κανονισμό για τα δεδομένα. Γιατί πρόκειται για 28 διαφορετικέ ένωμε τάξει που έχουν διαφορετικά πρότυπα εδώ στην Ένωση. Άρα να προσαρμοστούμε στα ισχύοντα και εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δούμε τι θα γίνει με την προστασία των δεδομένων και για στην περίπτωση της καταπολέμησης του εγκλήματος. Πιστεύω δε ότι καμία χώρα, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν το, δεν έχουν το περιθώριο να σέβονται τα ανθρωπίνα δικαιώματα που είναι κάτι τόσο σημαντικό. Ο μεγάλος αδερφός δεν πρέπει ούτε Γερμανός ούτε Αμερικανός. Ο επόμενος, δύο λεπτά. Μωράες. Α, γιατί συζητούμε αυτό το θέμα σήμερα. Αυτή η ερώτηση ετέθη, είμαστε σαφέστατοι. Μετά τις βασανιστικές έρευνες της NSA, ακόμα και είπα, ξεκίνησαν ένα ταξίδι διεθνών προδιαγραφών κατά της οικονομικής κατασκοπίας και προς προστασίας των πολιτών κατά της κατασκοπίας που δεν χρειάζεται καθόλου. Κατασκοπία κατά των τρομοκρατών για ανάγκες, πραγματικές ανάγκες ασφαλείας είναι κάτι σημαντικό. Αλλά όπως είπε και ο Επίτροπος, όταν μιλάμε για εταιρείες στη Δυτική Ευρώπη και ενδεχόμενες παραβιάσεις του γερμανικού και ευρωπαϊκού δικαίου, όπως σε αυτή την περίπτωση, τι συζητάμε, περί τίνος πρόκειται. Όπως είπε το The Spiegel και το Washington Post, ε, μια πολύ μεγάλη συμφωνία πραγματικά. Ε, δύο από τα μεγάλα κράτη-μέλη μας, Γερμανία και Γαλλία. Κάτι πολύ σημαντικό. Δεν θέλω να αναφέρω ξεχωριστά κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να αντιμετωπίσω και τη χώρα μου όσον αφορά την έρευνα για το NSA. Θα πρέπει εδώ σαν Κοινοβούλιο να ασχοληθούμε με την προστασία των πολιτών κατά ε, μη παραβίαση παραβίασης του ζωής. Και αυτό κάνουμε σήμερα. Ασχολούμεθα με εικασίες, πολλές κατηγορίες και εικασίες. Αλλά είναι σημαντικές όπως λέει η Washington Post και η Der Spiegel. Και τι πρέπει να κάνουμε. Να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε διαδικασίες εποπτείας. Δεν έχουμε αρμοδιότητες εδώ, αλλά όπως είπαμε και στην έρευνα για την NSA, θα πρέπει να ζητήσουμε από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν εκεί και δεν το κάνουν. Και εμείς σήμερα θα τους υπενθυμίσουμε. Πρέπει να ζητήσουν τα κράτη-μέλη να κάνουν συγκεκριμένα βήματα και να υπενθυμίσω σε κάποιους ότι η Bundestag της Γερμανίας έκανε πρόοδο εδώ, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι. Ένα, οι βουλευτές προσπάθησαν να προχωρήσουν και να αποκαλύψουν πολλά από αυτά. Καλά έκαναν και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν δικαίωμα να το κάνουν αυτό όταν απειλούνται τα θεμελιώδη δικαιώματα και το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ευχαριστώ. Για δύο λεπτά. Ο κύριος Βάιντεν Ευχαριστώ πρόεδρε. Πολύ φοβάμαι ότι δεν θα είναι η τελευταία φορά που θα ασχοληθούμε εδώ με τέτοια ζητήματα. οι μυστικές υπηρεσίες ε, λειτουργούν στο σκοτάδι και το σκοτάδι προκαλεί φόβο σε πολλούς ανθρώπους. Εμείς ως Κοινοβούλιο θέλουμε στην Ευρώπη της ελευθερίας, την ασφάλεια ε, να ζούμε. Και είναι λοιπόν ε, ένα δυνατό σημείο του κρατου δικαίου το γεγονό ότι οι αρμόδιοτητε τη αστυνομία και των μυστικών υπηρεσιών ορίζονται με σαφήνεια. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει δικαιολόγηση κάθε μέτρου και κάθε δράση και δεν θα πρέπει να υπάρχει συστηματική δράση. Τι χρειαζόμαστε λοιπόν, χρειαζόμαστε κοινοβουλευτικό έλεγχο, είναι καλό αυτό που κάνουμε εδώ, χρειαζόμαστε εντατικέ έρευνε σε όλη την Ευρώπη, σε όλα τα κρατημέλη όπου συμβαίνουν αυτά. Επίση χρειαζόμαστε ε, ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης ε, της ε, προστασίας των δεδομένων χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ασφάλεια στην Ευρώπη για να υπάρχει μια ευρωπαϊκή υποδομή και νομικό πλαίσιο για το ευρωπαϊκό νέφος. Κατά τέταρτον χρειαζόμαστε προστασία για τους πληροφοριδότες όπως ο Σνόντεν. Επίσης, κατά πέμπτον, χρειαζόμαστε Μία συμφωνία, διμερείς, ε, οι διμερείς συμφωνίες δεν έχουν προφανώς αξία. Χρειαζόμαστε λοιπόν ε, δέσμευση από όλα τα κρατημέλη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην υπάρχει επιχειρηματική κατασκοπία και κατά έκτον χρειάζεται τόλμη και θάρρος να ελέγξουμε τις διεθνείς συμφωνίες που έχουμε προσυπογράψει από το SWIFT. Θα πρέπει να τις εξετάσουμε και να ληφθούν σαφείς αποφάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξεγάγει τα συμπεράσματα από τις αποφάσεις μας και πιστεύω αξιότιμοι συνάδελφοι, αξιότιμοι υπέτροπε, ότι η ελεύθερη κοινωνία διακρίνεται από το γεγονός ότι είναι αντιτεθειμένη να ερευνήσει περιπτώσεις καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς να είναι αντιτεθειμένη να τις δεχτεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. ομιλητής, ο κύριο Γιάκοβιτ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στις... Ε, ε, κοινοβουλευτικές συζητήσεις, μιλάμε για τον τύπο, για πληροφορίες που προκύπτουν από τον τύπο. Φυσικά εδώ υπάρχουν πάρα πολλές αμφιβολίες και πάρα πολλές ενδείξεις. Αυτό είναι σαφές. Ακούσαμε επίσης ιδιαιτέρους ότι δεν έχει νόημα αυτή η συζήτηση. Αντιθέτως, έχει, έχει νόημα αυτή η συζήτηση και θα πρέπει να υποστηριχθεί το Γερμανικό Κοινοβούλιο προκειμένου να ελέγξει τα όλα όσα συνέβησαν. Να περάσουν όλα αυτά από ενταλλαχή έλεγχο. Αυτό που χρειαζόμαστε στην ε, Ευρώπη είναι μια πολυμερή συμφωνία. Δεν μπορούμε πραγματικά να επιτρέψουμε αμοιβαία κατασκοπία και θα πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη των πολιτών, εμπιστοσύνη των ε, θεσμών. Προκειμένου με τον τρόπο αυτό οι πολίτες και το πολιτικό σύστημά μας να προστατευτούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο παίρνει η Επιτροπός Γύρωβα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση αυτή που πραγματικά συμφωνώ ότι έχει νόημα και είναι πολύ καλό το, το, το ζήτημα αυτό εδώ τα εισαγωγικά μου σχόλια ήταν μάλλον μετριοπαθή και στεγνά, γιατί είπα ότι δεν έχουμε επαρκή αποδεκτικά στοιχεία και δεν έχουμε αρκετά τεκμήρια, μόνο κάποιες αναφορές του τύπου. Άρα, ως εκ τούτου, για μένα, ως ε, νομικό, είναι αδύνατον να εξαγαγώ συμπεράσματα ή να μην εξαγαγώ συμπεράσματα. Επίσης, μίλησα για την έλλειψη ευρωπαϊκής αρμοδιότητας, γιατί είναι θέμα στην αρμοδιότητα των κρατών μελών. Ωστόσο, θα πρέπει να σας πω ότι μετά από αυτά που άκουσα για τι πληροφορίε για τα υποτιθέμενα καινούργια σκάνδαλα για την κατάχρηση των ε, δεδομένων από την NSA. Ε, είμαι σε νέο καθεστώς επαγρύπνησης, γιατί είμαστε σε μια φάση, όπως ξέρετε, διαπραγματεύσεων με τις Αμερικανικές Αρχές. Mm για το σύστημα του ασφαλούς λιμένα, το Safe Harbor, όπου διαπραγματευόμαστε τις εξαιρέσεις υπό τις οποίες οι μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα των Ευρωπαίων πολιτών ή των ε, νομικών προσώπων που επισέρχονται στο σύστημα των ΙΠΑ. Ε, Αυτό δεν πρόκειται να διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις σας. Διαβεβαιώ η ε, ευάλωτη και ευαίσθητη εμπιστοσύνη που έχουμε πετύχει δεν θα ωφεληθεί. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση α, ακούγοντας αυτό το έχουμε ακούσει τις ειδήσει αυτές. Είμαστε σκληροί στις διαπραγματεύσεις. Θέλουμε να δούμε τους κανόνες, τις αρμοδιότητες που ισχύουν από αμερικανικής πλευράς, αλλά επίσης θέλουμε να λάβουμε συγκεκριμένες ε, ασφαλιστικές δικλείδες από πλευρά της Αμερικανικής ε, κυβέρνησης για το ότι θα ακολουθηθούν οι κανόνες αυτές. Άλλο λοιπόν ε, είναι οι κανόνες, γραπτοί οι κανόνες και άλλο είναι η εκτέλεση των κανόνων αυτών. Επαναλαμβάνω, είναι σκληρές οι διαπραγματεύσεις αυτές και αυτό θα σημαντέψει τις επόμενες εβδομάδες. Καθότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις μέχρι τα τέλη του Μαΐου για να πετύχουμε συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένες, συγκεκριμένους κανόνες στα πλαίσια του Safe Harbor. Να σας ενημερώσω λοιπόν ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι σε εξέλιξη, συνεχίζονται και επίσης παράλληλη διαδικασία είναι η διαδικασία όρις, ε, ε ολοκλήρωσης της ε, κανονισμού για την προστασία των δεδομένων. Μαζί με την οδηγία για την αστυνομία. Αυτό για να λάβετε τις πιο πρόσφατες ε, ειδήσει για το τι συμβαίνει στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. Ε, ολοκληρώθηκε λοιπόν αυτή η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη και καθώς αλλάζουμε από πλευρά τη Επιτροπή των Εκπρόσωπων να ζητήσουμε από τον Επιτροπό Χίλ να κάτσει στη θέση του και συνεχίζουμε τη συζήτηση. Να δώσω το λόγο στην ε, εισηγητρία την κυρία Γκίλη, η οποία και έχει πέντε λεπτά.